Ladies and Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και φίλοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω εδώ στο Κοινοβούλιο. Ίσως μερικοί έρχεστε και για πρώτη φορά. Πράγματι. Ε, ναι, ναι, βλέπω, το βλέπω. Υπάρχουν και άλλοι ευρωβουλευτές Χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν είμαι μόνος μου εδώ για να παρουσιάσω το, Ευρωπαϊκό, το βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Δημοσιογραφία. Καταρχάς, όλοι κερδίσατε γιατί όλοι σας είστε εθνικοί νικητές και βραβευμένοι και γι' αυτό η κριτική επιτροπή είχε πολύ δύσκολο έργο να επιλέξει μεταξύ των καλυτέρων. Τέσσερις. Πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα για τρίτη φορά απονέμεται το βραβείο του καλύτερου δημοσιογράφου. Και ακόμη πιο σημαντικό αναγνωρίζουμε τα εξαιρετικά επιτεύγματα των δημοσιογράφων και καλωσορίζω ιδιαίτερα τους νέους δημοσιογράφους διότι έχουμε οργανώσει το εργαστήριο που φέρει τον τίτλο «Δημοσιογράφη είδος σε κίνδυνο» με ερωτηματικό. Εδώ και ένα χρόνο είχαμε αποφασίσει να κάνουμε την απομονωμή για το 2009, πολύ σημαντικό έτος για το Κοινοβούλιο γιατί άρχισε να ισχύει πριν από ένα χρόνο η συνθήκη της Λισαβόνας μετά από τα προβλήματα που συνάντησαν ορισμένες χώρες μέλη που δεν θα τις αναφέρω εδώ. Και χρειάστηκε να ανταποκριθούμε στην κρίση, στην χρηματοπιστωτική κρίση μέσω νομοθεσία, τη στρατηγική του 2020, δομικές μεταρρυθμίσεις που σε μερικές χώρες μόλις αρχίζουν πάρα πολύ σκληρά μέτρα για μερικές χώρες και επίση θέλουμε να εφαρμόσουμε μια στρατηγική εξόδου από την κρίση για να αποφευχθεί η αποτελμάτωση που άρχισε να σημειώνεται και στη δεκαετία του 30 του προηγούμενου αιώνα μετά την κρίση. Η κάλυψη των δημοσιογράφων πρέπει να είναι φυσικά ανεξάρτητη και ουδέτερη και είναι ουσιώδης προϋπόθεση για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πανενωσιακή συζήτηση στον δημόσιο χώρο. Με τη δημιουργία του βραβείου αυτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προωθήσει κριτικό και αμερόληπτη, κριτική και αμερόληπτη δημοσιογραφία. Όλοι μας και οι 736 αναγνωρίζουμε το θάρρος σας. Θέλουμε πραγματικά αμερόληπτη και κριτική δημοσιογραφία και γι' αυτό Γνωρίζω βέβαια πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσετε στο κοινό την πολιτική της Ένωσης πράγμα πάρα πολύ πολύπλοκο μερικές φορές και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να καταστούν όλα αυτά ενδιαφέροντα για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες θέλουν να διαβάζουν κάτι ενδιαφέρον αλλά μερικοί πολιτικοί δεν θέλουν να φύγονται πολύ αμφιλεγόμενα θέματα, αλλά αφού υπάρχει ανταγωνισμός παντού, φυσικό είναι αυτό. Μερικοί πολιτικοί κατηγορούν, ψέγουν τα μέσα ενημέρωσης ότι δεν είναι αντικειμενικά, αλλά θα ήθελα να ξανατονίσω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο να παρουσιάσει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες απλά. Τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων το ξέρουν αυτό καλά και εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου για 50 σχεδόν χρόνια η δημοσιογραφία δεν είχε το δικαίωμα να δημοσιεύει αυτά που πίστευε και να εκφράζει με παρησία αυτά που αισθανόταν. Ξέρω λοιπόν καλά πόσο πολύτιμες είναι οι ενωσιακές αξίες. Πριν από 25-30 χρόνια σε πολλές από τις χώρες μας δεν ήταν εύκολη η δουλειά σας. Και πιστεύω ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό να επενέσουμε όσους επικρίνουν την πολιτική μας γιατί μας αναγκάζουν να τη βελτιώσουμε και καμιά φορά δείχνουν τα λάθη που μπορεί να έχουμε κάνει. Λένε ότι οι πολιτικοί παραπονούνται για τα μέσα όπως η γεωργοί για τον καιρό ή η ναυτική για τη φουρτούνα. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε στις επαφές μας και στις επικρίσεις μας κατά των μέσων. Εσείς τα ξέρετε βέβαια. Και στη δική μου χώρα χρειάστηκαν πολύ σκληρές μεταρρυθμίσεις επί τέσσερα χρόνια. Αλλά ήταν μεγάλο στήριγμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην προσπάθεια αυτή των μεταρρυθμίσεων γιατί είναι πάντα δύσκολο για τους πολίτες, πάντοτε δύσκολο να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις και είναι και δική σας ευθύνη να καταλάβετε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι πάντοτε δύσκολη κατάσταση. Αλλά σε δύο, τρία, τέσσερα χρόνια έρχεται η νίκη και θα ήθελα να το γνωρίζετε όλοι. Είναι κοινή μας ευθύνη πολιτικών και δημοσιογράφων να καταλαβαίνουμε όχι μόνο το σήμερα αλλά και το αύριο και το μεθαύριο. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στην απονομή, θέλω πρώτα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του βραβείου, εσάς τους δημοσιογράφους στις χώρες μέλη που συμμετέσχατε και που πήρα το γενικά μέρος και τα μέλη και των Εθνικών Κριτικών Επιτροπών και της Κριτικής Επιτροπής των Βρυξελών που διάβασε, παρακολούθησε, άκουσε και αποτίμησε πλήρως και προσεκτικά όλες τις υποψηφιότητες στον ελεύθερο μάλιστα χρόνο της. Ευχαριστώ επίσης την Αντιπρόεδρο κυρία Ρώδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου που προείδρευε της Επιτροπής, την κυρία Μέρι Χόνιμπολ και τον Ζαν Μαρίκα Καβαντά που ήταν μέλη της. Ο συνάδελφος Βίλαντ επίσης είναι εδώ, Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, όπως και η κυρία Ρώδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο συνάδελφος Ζαν Καβαντά. Όχι, όχι, όχι. Η Μαρία Χόνιμπολ και εκείνο εργάστηκαν πολύ σκληρά. Αλλά και δημοσιογράφοι. Ιδιαίτερα ο κ. Λορέντσο Κονσόλη. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Γουανέλα Χος που η δική της διεύθυνση ήταν υπεύθυνη για την απονομή. Και τώρα, και τώρα να τελειώσω. Κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα, ούτε εγώ δεν το ξέρω. Ξέρω μόνο ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες. Γραπτός τύπος, ίντερνετ, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Αρχίζουμε λοιπόν. γραπτός τύπος. Πρώτον, ο γραπτός τύπος. Η παρουσία των δημοσιογράφων σε θέματα της παράνομης μετανάστευσης, πρόβλημα που ακόμη δεν έχει επιληθεί η Επιτροπή επέλεξε συνενετικά ένα άρθρο που το θεώρησε εξαιρετικό και με μεγάλη δημοσιογραφική αξία και όπως είπε ένα μέλος της Επιτροπής η ανάγνωση του άρθρου αυτού ήταν σαν να διάβαζε κανείς λαγατεχνία και το βραβείο απονέμεται στον Βίτολντ Σαμπρόσκι από την Πολωνία. Για το άρθρο σήμερα θα εκβραστούν δύο πτώματα. Το άρθρο δημοσιεύτηκε από την Γκαζέτα Βιμπόρτσα. Πρώτη φορά έρχεστε στο κοινοβούλιο. Μάλιστα.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 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να ζητήσω συγνώμη από τους συναδέλφους που ήρθαν εδώ γιατί πήρα εγώ το βραβείο. Και δεύτερον, διότι θα ήθελα να πω μερικά πράγματα στη γλώσσα μου, ελπίζω να το κατανοείτε αυτό. Είναι δύσκολο να μιλάει κανείς αγγλικά σε τέτοιες στιγμές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είμαι σίγουρος ότι εσείς θα τα καταφέρετε να καταλάβετε. Κυρίες και κύριοι, είμαι βαθιά συγκινημένος, είναι προφανές αυτό. Και είμαι επίσης βαθιά συγκινημένος διότι, όπως είπε ο Πρόεδρος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά την κριτική σκέψη των δημοσιογράφων και το γεγονός ότι επιβραβεύθηκε το άρθρο μου σημαίνει ότι πράγματι το Κοινοβούλιο εκτιμά την κριτική δημοσιογραφία. Το κείμενο ήταν σημαντικό για μένα, για προσωπικούς λόγους. Πρώτα ως Πολωνός που ζει σε μια χώρα η οποία κάποτε απέστελε σε όλο τον κόσμο τεράστια κύματα παράνομων μεταναστών σήμερα ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορώ, κατάφερα να πάω, μπόρεσα να πάω στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος και να δω τις μικρές βαρκούλες με τις οποίες προσπαθούσαν οι άνθρωποι να περάσουν το ποτάμι. Μερικοί από αυτούς καταφέρνουν να επιβιώσουν, να φτάσουν, μερικοί όχι και χάνονται. Όλο και λιγότεροι καταφέρνουν να φτάσουν σε κάποιο αίσιο πέρας ας πούμε της προσπάθειάς τους. Οι άνθρωποι αυτοί μου θύμισαν τους ανθρώπους που γνώριζαν, που γνώριζα εγώ μάλλον, όταν ζούσαμε ακόμα υπό κομμουνιστικό καθεστώς και οι άνθρωποι αυτοί εγκατέλειπαν την Πολωνία που ήταν εξαιρετικά πτωχή χώρα τότε για να πάνε αλλού να ζητήσουν την τύχη τους. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω το βραβείο αυτό σε όλους αυτούς τους φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι, δύο έγραψα το άρθρο. Uh, Τώρα θα ήθελα να πω μερικά λόγια για τον συνάδελφο Γκάλαγκερ και Γκάλι που ήρθαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ, τους. Να τους ευχαριστήσω και αυτούς δηλαδή, γιατί μαζί τα οργανώσαμε όλα, όλοι οι ευρωβουλευτές. Δεύτερη κατηγορία, ίντερνετ Πρόκειται για ένα blog από το Ηνωμένο Βασίλειο και ο συγγραφέας γράφει υπό το ψευδόνυμο Nose Monkey. Το άρθρο του αφορά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ένωσης, τι ποσοστό της εθνικής νομοθεσίας προέρχεται από την Ένωση. Σύμφωνα με την Κριτική Επιτροπή, ο συγγραφέας έχει κάνει πολύ μεγάλη ερευνητική δουλειά, το άρθρο του είναι ευνόητο, πιστικό και χιουμοριστικό. Έχει κάνει πολύ στατιστική και αναλυτική δουλειά και συγκρίσεις. Ταυτόχρονα όμως το άρθρο του διαβάζεται με μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι και αυτό σημαντικό. Επιστημονική δουλειά και πολύ ευχάριστο άρθρο. Και εγώ ήμουν επιστήμονας και ξέρω πόσο δύσκολος είναι ο συνδυασμός. Λοιπόν, τον συγχαίρω. το βραβείο αποδίδεται στον James Clive Matthews από το Ηνωμένο Βασίλειο για το άρθρο «Τι ποσοστό της νομοθεσίας προέρχεται από την Ένωση». Φυσικά σας δίνουμε το λόγο, αλλά αναμένουμε και την ακριβή απάντηση. Θα είμαι σύντομος. γιατί χθε πήγα σε κάποιο είδο κάποιο είδος δεξίωση ενό λόμπι. Καταλαβαίνετε τέλο πάντων. Ε, πήγα μέχρι αργά. Ε, ναι, κατανάλωσα πολύ. Πάνω από 50% λέει ο πρόεδρο. Ναι, μάλλον. μάλλον κάπου εκεί, κάπου εκεί. Ε, ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τηλεόραση 2010. τηλεόραση. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα Euphoria παρουσιάζει την ιστορία της Ένωσης με εύληπτο και διασκεδαστικό τρόπο για τους νεότερους. Το πρόγραμμα αποτελεί τεράστιο όγκο πληροφόρησης και χρησιμοποιεί συναισθηματικούς τρόπους επικοινωνίας. Η Κριτική Επιτροπή επένεσε ιδιαίτερα τη φαντασία των δημοσιογράφων που είναι σημαντικό στοιχείο για τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι ελκυστικό, διασκεδαστικό και επιμορφωτικό ταυτόχρονα. Και ο νικητής είναι ο Νέμετ Σόλτ από την Ουγγαρία για το πρόγραμμα Euphoria Νέμετ Σόλτ. And this program... Το πρόγραμμα εξέπεμψε η MTV. Λέγομαι Ζολτ Νέμετ, είμαι Ούγγρος πολίτης. Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο αίσθημα της ευρωπαϊκής κοινότητας, αλλά ελπίζω να είχα. Έτσι αρχίζει, με αυτά τα λόγια αρχίζει το φιλμ, η ταινία αυτή, που ξεκίνησε από την εντύπωση, από την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακριά από τον Ούγγρο πολίτη. Παρόλες τις διάφορες ε, προμοσιών, παρόλα τα, ε, τις ειδήσεις, τα ραδιόφωνα κτλ. Δεν, έχουν ακούσει, δεν έχει ακούσει ο μέσος Ούγγρος τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλησα λοιπόν να τους εξηγήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο διαφορετικό. Ήθελα να πω με απλό και διασκεδαστικό τρόπο τι είναι. Ήθελα να προσελκύσω την προσοχή των συμπολιτών μου, ιδίως της νεότερης γενεάς. Το μέλλον των νέων γενεών ταυτίζεται στο μέλλον όλης της ευρωπαϊκής κοινότητας. Η προσοχή της νεότερης γενεάς μπορεί να προσελκυστεί μόνο με τρόπο διασκεδαστικό παιχνιδιάρικο. Θέλαμε να φτιάξουμε λοιπόν ένα επιμορφωτικό ε, ντοκιμαντέρ, μια επιμορφωτική ταινία που να είναι διασκεδαστική, να είναι κατανοητή χωρίς μεγάλη προσπάθεια, να προσπαθεί να εξηγήσει την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι με τρόπο διδακτικό αλλά με τρόπο ε, σαν να είναι παιχνίδι. Να προσελκύσουμε λοιπόν την προσοχή των ε, προσώπων αυτών και όποιος ενδιαφέρεται περισσότερο μπορεί να βρει και άλλες ακριβέστερες πληροφορίες από το διαδίκτυο. Όταν λοιπόν φτιάξαμε την ταινία την δοκιμάσαμε. Οι νεαροί που την είδαν την εκτίμησαν πολύ. Είπαν ότι τους διευκρίνησε πολλά πράγματα η ταινία. Λίγοι όμως από αυτούς θέλουν να γίνουν εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τελείωσε η ταινία είχα μια ιδέα. Θέλησα να το αντιγράψω και να στείλω πολλά αντίγραφα σε σχολεία και να μπουν στα μαθήματα. Πήραμε την ταινία και στο Στρασβούργο και την δείξαμε σε ορισμένους εμπειρογνώμονες. Προσπαθήσαμε να ε, λάβουμε και κάποια επιδότηση για να φτιάξουμε τις κόπιες, αλλά δεν κατάλαβαν για ποιο λόγο ήταν τόσο σημαντικό για μας. Ίσως να φταίω εγώ. Ίσως έπρεπε να είχα, εξι, να είχα ε, επιλέξει μια άλλη πόλη για την προσπάθεια μου αυτή. Ίσως τις Βρυξέλλες. Σείς, κύριε Πρόεδρε και η Κριτική Επιτροπή κατανοήσατε την σημασία της ταινία. Εγώ πάντοτε εμπιστευόμουν την κρίση σας. Ήμουν βέβαιος ότι θα σημειώσω επιτυχία. Έτσι έγραψα λοιπόν την ομιλία μου από πριν για να μπορώ να τα διαβάσω γιατί δεν μιλώ καλά αγγλικά. Η ταινία μου λοιπόν κατέκτησε το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, δημοσιογραφία. Εσείς ε, κατανοήσατε καλά τι σημαίνει να μπορεί κανείς να εξηγήσει με απλό τρόπο τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με απλό και διασκεδαστικό τρόπο. χωρίς να μειώνει την αξία του περιεχομένου. Ίσως οι εμπειρογνώμονες να την εκτιμήσουν αυτή τη φορά, μετά την βράβευση δηλαδή. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι, τελειώνουν τα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου. Το βραβείο δεν ανήκει μόνο σε μένα, το βραβείο ανήκει και στους συναδέλφους μου που εργάστηκαν στην Ουγγαρία στο περιφερειακό στούντιο της Ουγγρικής τηλεόρασης. Το βραβείο δείχνει εν τέλει ότι μπορεί να είναι σημαντική η παραγωγή όχι μόνο στις πρωτεύουσες των κρατών αλλά και στις περιφέρειες. Εσείς με το βραβείο βραβεύετε όχι μόνο εμένα αλλά και την Ουγγρική τηλεόραση. Αναγνωρίζετε ότι η τηλεόραση αυτή μπορεί να παραγάγει αξιόλογα προγράμματα. Η επόμενη Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η Ουγγρική. Οι συνάδελφοί μου και εγώ είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε το καθήκον μας στην Ουγγρική τηλεόραση. Εγώ είχα ήδη ένα αίσθημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Είναι, δεν είναι τίποτα, είναι κάτι τεχνικές διευκρινήσεις. Λοιπόν, τέταρτη κατηγορία. Τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντική. Το ραδιόφωνο 2010 και αυτό. Ραδιόφωνο. Πρόκειται για μία έρευνα που δείχνει ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση δεν φτάνει πάντοτε στους αγρότες the στην Τουρκία. Σύμφωνα με την Κριτική Επιτροπή, οι δημοσιογράφοι διάλεξαν πολύ καλό θέμα. Έκαναν εξαιρετική έρευνα και στην τουρκική Ήπεθρο και στην Άγκυρα. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επένεσαν την τέλεια διάρκεια και τη χρονική στιγμή στην οποία εξεπέμφθη το πρόγραμμα γιατί κράτησε ζωντανή την προσοχή των ακροατών. Τώρα λοιπόν το βραβείο ραδιοφωνίας Κάσια Νόρελ και Νούρι Κίνο από τη Σουηδία για την χρηματική στήριξη της Τουρκίας από την Ένωση. Ορίστε κυρία μου και κύριε. Το πρόγραμμα εξεπέμφθη από το Σουηδικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Έκολτ. Θα χρειαζόταν εδώ μια γυναίκα, αλλά δυστυχώς είναι στην Αυστραλία. Α, στην Αυστραλία. Α, μάλιστα. Well, um Όπως είπα, δυστυχώς η Αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφος δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Όταν γινόταν η παραγωγή ε, ήταν ήδη στον ένα το μήνα της εγκυμοσύνης για το δεύτερο παιδί της. Και δούλευε μάλιστα και από, την, ε, από το νοσοκομείο, από την κλινική δηλαδή. Θα ήθελα λοιπόν να μεταφέρω τις ευχαριστίες μου στο σουηδικό ραδιόφωνο και στη Σεσίλια Ρούς που ε, τα κατέστησε δυνατά αυτά, που πίστεψε σε εμά, μας έδωσε την ε, δυνατότητα να, ε, και μας δίνει τη δυνατότητα να ψάξουμε να βρούμε τις διάφορες οικονομικές ανομαλίες σε όλο τον κόσμο. αυτό το πολύτιμο βραβείο βραβεύει κυρίως τις πηγές μας, τους αγρότες, τις γυναίκες στην Ανατολική Τουρκία Επίσης, στους συναδέλφους μας ολόκληρου του κόσμου που εργάζονται υπό όλο και δυσμενέστερες συνθήκες. Βραβεύεται τους ανθρώπους που βρίσκονται στις φυλακές και τους δημοσιογράφους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους πράττοντας το καθήκον τους. Το καθήκον τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη η χαρά μας που δίνουμε τα τέσσερα αυτά βραβεία. Αλλά σας βεβαιώνω ότι για μας όλοι είστε νικητές. Είστε περίπου 100 από τις 27 χώρες μέλη, χωρισμένοι σε τέσσερις κατηγορίες. Νικητές στις εθνικές κατηγορίες σας, στους εθνικούς διαγωνισμούς σας. Και είναι πολύ δύσκολο να επιλέξει κανείς τον άριστο μεταξύ των αρίστων. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβετε και μας, αλλά πρώτα πρώτα συγχαρητήρια στους τέσσερις νικητές που κάθονται εδώ μεταξύ μας και θα ακολουθήσει το επόμενο βραβείο σε ένα χρόνο αλλά θέλαμε να σας προσφέρουμε και μια μικρή έκπληξη ίσως είναι και μεγάλη έκπληξη προ μόνο σε συνεργασία με το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γι' αυτό και το μικρό διάλειμμα που έκανα πριν, την επίσκεψή σας όπου θέλετε, απανταχού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν επιθυμεί κάποιος από εσά και δεν γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κτίρια μας, τον τρόπο που εργαζόμαστε, είναι σημερινή. Η σημερινή μέρα είναι εργάσιμη μέρα. Κάθε μέρα είναι εργάσιμη μέρα. 70% νομίζω όπως είπε κάποιος από τους σας προηγουμένως προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, της Εθνικής Νομοθεσίας δηλαδή. Δεν κάνουμε πάντοτε έξοχη εργασία, κανείς δεν είναι τέλειος. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα μας κρίνεται και θα μας επικρίνεται. Από καιρό σε καιρό χρειαζόμαστε βέβαια και κανένα θετικό άρθρο Καλά θα ήταν να πείτε κάτι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους ευρωβουλευτές. Σήμερα θα σας δείξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εκπρόσωπος της διοίκησής μας, είναι εκπρόσωποι όλοι, κάθονται εδώ. Στο τέλος της ε, συνάντησής μας μπορείτε να έλθετε εδώ και να οργανωθείτε. Όλα γίνονται στο άψε σβήσε, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν είχε προγραμματιστεί αλλά είναι ε, θαυμάσια η ατμόσφαιρα εδώ και είμαστε ευγνώμονες σε όλους και όλες που ήρθατε εδώ. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας και θα σας δω ξανά του χρόνου. Well, well, it's a good idea. And now... Άλλη μια θαυμάσια ιδέα. Όλοι εδώ λοιπόν ας έλθουμε εδώ και θα βγάλουμε φωτογραφίες. Ο φωτογράφος θα σταθεί πάνω στο έδρανο. Όλοι ελάτε εδώ. Σε δύο, τρεις σειρές, τέσσερις, όσες θέλετε. Ο φωτογράφος να ανέβει στο τραπέζι. Okay. Young journalist, young... Οι νεαροί δημοσιογράφοι, οι νεαροί. Να οργανωθείτε.